Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας με το σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη, ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες με την εισηγήτρια κυρία Σόιντροβα. Το λόγο έχει η ίδια η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή εξετάζει την ισότητα ανδρών και γυναικών στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η τέταρτη εξουσία τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Επηρεάζουν ιδιαίτερο στην κοινωνία μας, τα πολιτικά πράγματα. Γι' αυτό ζητήσαμε από ανεξάρτητο ε, οργανισμό να διεξαγάγει μελέτη για το τι συμβαίνει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ε, κοιτάξαμε λοιπόν το κατά πόσον υπάρχει διακριτική μεταχείριση και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις πολλές καλές τροπολογίες στην έκθεσή μου. Καμιά εκατοστή. Ευχαριστώ λοιπόν για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό. Επεξεργαζόμαστε συμβαστικέ λύσεις και ελπίζω ότι θα γίνουν ε, γενικώ αποδεκτές κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Στις συμβιβαστικές μας προτάσεις μελετήσαμε το κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση των γυναικών στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κατά τα άλλα πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα και την ανεξαρτησία των μέσων η δική μου προσέγγιση είναι να ενθαρρύνουμε τα θεσμικά όργανα των κατόμελων και τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και να δείξουν περισσότερη ευαισθησία στην ισότητα των φύλων, στην προβολή τους στα μέσα. Ε, η εικόνα των γυναικών στις διαφημίσεις και στα μέσα θα πρέπει να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μην χρησιμοποιεί σεξιστικά πρότυπα και άλλα στερεότυπα σεξιστικά. Ε, θα πρέπει να δοθούν ε, κατάλληλα εκπαιδευτικά παραδείγματα, ε, τα οποία ε, μέσα από την, τον εκπαιδευτικό τομέα θα είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικά από άλλα αποτρεπτικά μέτρα. Γι' αυτό δεσμευτικέ ποσοστώσει, ποινέ, επιβολή προστήμων ή οτιδήποτε άλλο δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. Λόγω χάρη για το σεξισμό στη διαφήμιση. Είναι αρμοδιότητα των 100 μελών αυτά. Όμω κάποια ζητήματα πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Δηλαδή η βία κατά των γυναικών και η παρενόχληση. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας υποτίθεται ότι εξυπηρετούν την κοινωνία συνολικά. Η δομή τους και η δουλειά τους θα πρέπει να κατατοπίζουν το γεγονός ότι η γυναίκα είναι το ίμιση του πληθυσμού της κοινωνίας η εξέβρεση εργασία είναι δύσκολη και από τη σκοπιά τη εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε περισσότερο εδώ και να βεβαιωθούμε ότι οι ευθύνε που αναλαμβάνουν και σε τομεί ε, διοίκηση στα μέσα μαζική ενημέρωση είναι μεγαλύτερε. Ε, η μελέτη θα ε, παρουσιαστεί από την Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων σε λίγα λεπτά. Ελπίζω στη συνεργασία σας και στο εγγύς μέλλον και ελπίζω ότι θα είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη συζήτηση στην Επιτροπή μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Σόιντροβα και τώρα ο λόγος του σκιώδης εισηγητές, η κυρία Λιλιάνα Ροντρίγκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για την ισότητα των φίλων στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι καθοριστική σημασίας θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντας τη δημοσιογράφο του BBC, η οποία ε, δούλεψε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας πάνω από 30 χρόνια και λόγω της μισθολογικής διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών εγκατέλειψε τη θέση της ε, ως ανταποκρίτρια του BBC στην Κίνα. Πέρσι αποκαλύφθηκε από την BBC ε, ο μισθός ε, των ανωτέρων στελεχών της και η ίδια δημοσιογράφος έδειξε ότι υπάρχει αναντήρητα μισθολογικό χάσμα μεταξύ άνδρων και γυναικών που κάνουν την ίδια δουλειά. Πάνω από 200 υπάλληλοι της BBC υπέβαλαν ε, προσφυγή ζητώντας να διορθωθεί το μισθολογικό χάσμα και να δοθεί ίση αξία σε άνδρες και γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά. Έτσι βλέπουμε ότι ο το BBC που είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται από δημόσιο χρήμα ε, αναγνώρισε ήδη αναγκαστικά την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν τα ε, διάφορα κράτη-μέλη να παρακολουθήσουν το τι συμβαίνει στα δικά τους μέσα και ο καθένα να αναλάβει τι ευθύνε του, ιδίω στην περίπτωση δημόσιων υπηρεσιών. Ε, θέλουμε μια κοινωνία ισόρροπη και σωστά δομημένη. Θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα και για τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιες ε, βασικές αξίες θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και στην ε, σύνταξη τη έκθεση που τώρα συζητάμε. Η αναφορά στην ανισότητα των φύλων παραμένει στην ιεράρχηση των διάφορων ε, κλιμακίων των στελεχών ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα της ποσόστοσης σε ευρωπαϊκά, ε, δημόσια και κρατικά, μαλοκρατικά και ιδιωτικά δίκτυα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της εκπροσώπησης στην κοινωνία με στερεότυπα των, διαφόρων, των δύο ισότητα των φύλων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες και στις ε, ευκαιρίες σταδιοδρομίας και στην ε, προβολή των δύο φύλων ε, στα δίκτυα. Δεν θα πρέπει να μας δυσκολεύει ούτε καν επιβολή προστήμων και να θα μπορούσαμε να την προτείνουμε. Επίσης κάποιες συστέσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ανεξάρτητος που να ελέγχει το τι συμβαίνει. Επίσης οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι ενώσεις γυναικών και η ΛΟΑΔ θα πρέπει να μπορούν να συμμετάχουν στη σύνταξη αυτών των πολιτικών. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αρχές εξισορρόπησης επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική που να καταπολεμά τη σεξουαλική και ηθική παρενόχληση, να φροντίσουμε την σωστή προβολή των γυναικών στα μέσα θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και η συμπεριφορά στην κοινωνία με την ίδια λογική που το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει ότι περνάει από το χέρι του για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε, Λιλιάνε. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Μαρσελεζή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που χθε η Επιτροπή Απασχόλησης ψήφισε μια τόσο καλή έκθεση όπως τη δικιά μας. Γιατί εμείς εδώ πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και ξέρουμε ότι τα ΜΜΕ συμβάλλουν στην διαιώνιση αυτών των στερεοτύπων. Ήταν λοιπόν απαραίτητο να είχαμε μια ισχυρή και φιλόδοξη έκθεση, ώστε να κάνουμε κάποια βήματα παραπέρα, όπως πρέπει. Να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Η αυτορύθμιση καταρχάς, γιατί αυτό δεν φτάνει. Αν έφτανε η αυτορύθμιση δεν θα ήμασταν εδώ να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε έκκληση για δράση στι χώρες μέρη και στην Ένωση, από την οποία ζητάμε και από τα κράτη να κινηθούν και να δράσουν. Αυτό πρέπει να είναι τμήμα της έκθεσης και μπορεί να είναι αυτή με υπέρ. Να έχουμε δηλαδή μια πλειοψηφία εδώ στην Επιτροπή μας για θέματα διαφήμισης όπου βλέπουμε τα περισσότερα στερεότυπα και όπου πρέπει να παρανεύουμε περισσότερο για θέματα ισότητας. Επίσης υπάρχει υποεκπροσώπηση των γεγονών στην διεύθυνση και στη διοίκηση. Οπότε και πάλι πρέπει να επιμείνουμε ώστε να υπάρχει μια οδηγία που θα αφορά τα διοικητικά συμβούλια και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την ποσότητα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Έχουμε και άλλο ένα παλαιό αίτημα εδώ στην Επιτροπή μας, να έχουμε δηλαδή μια οδηγία για την γονική άδεια, Μητρική και πατρική, ώστε οι γονείς που είναι σε διοικητικές θέσεις να είναι σε θέση να διαχειριστούν και το χρόνο πατρότητας και μητρότητάς τους. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που συζητάμε εδώ στην Επιτροπή μας και νομίζω θα βρεθεί πλειοψηφία πέρα αυτών των ιδεών. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος επιθυμεί το λόγο. Η κυρία Σαντρόβα, εισηγήτρια, αφού όχι. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας και την προσέγγιση σας. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και θα βρούμε τους κατάλληλους συμβασμού όπου χρειάζεται. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και προσβλέπω στη συνέχιση των επαφών μας. Thank you. And now to the, uh, we are going to the next point on the agenda, study on gender. Επόμενο σημείο. Η κυρία Άννα Σίμονς. ερευνήτρια για αυτό το θέμα. Έχετε 20 λεπτά. 15-20 λεπτά. Okay, so yes, I'm, I'm here to uh, present our research. Uh, my name is Dr. Anna Fitzsimons from Opsit Research, and I'm here. Είμαι επιφορτισμένη με το θέμα της ότας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα ΜΜΕ. Ε, ορισμένες, ε, θα αναφερθώ μέσα από τις ε, δράσεις που αναλαμβάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε κάποιες συστάσεις για ανάληψη περαιτέρω δράσεων. Okay. Uh, so for this research, we review the existing literature. Να επισκοπήσουμε τις στατιστικές όσον αφορά το περιεχόμενο των ΜΜΕ όσον αφορά το, πολιτικό, το πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν ε, μελέτη στην Αυστρία, τη Μάλτα, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Χρησιμοποίησαμε 37 συνεντευξείς με γυναίκες που δουλεύουν στα μέσα και ε, με όσους δουλεύουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουν την ισότητα μεταξύ των γυναικών. Ε, τώρα, σε αυτά τα περιεχόμενα, οι γυναίκες εμφανίζονται σε έναν, με ένα στερεότυπο τρόπο, σε βοηθητικούς ρόλους, εστιάζοντας τον ρόλο τους στον οικοκυριό κλπ. Ε, έχουν, ε, είναι λιγότερο σοβαρές και έχουν μικρότερο, μικρότερη αυθεντία στην ε, δουλειά που κάνουν. Τώρα, όσον αφορά την ανισότητα στο προσωπικό των media, γίνονται διακρίσεις και οι περισσότερες από τις γυναίκες που έδωσαν συνεντεύξεις είπαν ότι υπάρχει μεγάλη ανισότητα, σοβαρές διακρίσεις βάρος του, σεξουαλική παρανεχόληση ε, και και ανισότητες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της παρουσίασης. Είχαμε και άλλα τεκμήρια για να δούμε τι γίνεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις ανισότητες που υπάρχουν σε σχέση με την πραγματικότητα των γυναικών. Ε, περιγράφονται πάρα πολλά παραδείγματα ε, γυναικών που παρουσιάζονται με έναν ε, υπεραπλουστευμένο τρόπο. Θα επανέλθω στα θέματα αυτά, αλλά πριν το κάνω θα ήθελα να θέσω ορισμένα από, τα, από τους τρόπους το πώς η ανισότητα ε, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και ποια είναι τα περιεχόμενά της. Ε, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα υπάρχει μεγάλη ποικιλία, πολυμορφία στις, στο επίπεδο των χωρών μελών, στο πώς προσλαμβάνονται οι ανισότητες μεταξύ των ε, φύλων. Αλλά ε, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έχουν γίνει σε εκείνες τις χώρες μέλη που έχουν υπερβεί το επίπεδο των ε, ποσοστώσεων. Στο δημόσιο χώρο οι οργανώσεις των ΜΜΕ ε, βρίσκονται σε καλή κατάσταση από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Παρ' όλα αυτά και εδώ υφίστανται σοβαρές διακρίσεις εις βάρος των γενικών που δουλεύουν για, σε δημόσια κανάλια, για παράδειγμα. Και υπογραμμίστηκε κατ' επανάληψη ότι ένας παράγων κλειδί, ο πιο σημαντικός, είναι το να έχει... Είναι το, το, ζήτημα των ε, ανώτερων θέσεων και δεν υπάρχει όμως σε κανένα κλάδο δεν υπάρχει η κατάσταση δεν είναι καλύτερη σε κανέναν απολύτως ε, κλάδο αλλά οι διακρίσεις αυτές είναι διαδεδομένες σε όλους τους ε, κλάδους. Ε, υπάρχει, υπάρχουν βέβαια κάποια χάσματα στην έρευνα τα οποία θα έπρεπε να πληρωθούν η εθνότητα, η ηλικία και το κοινωνικό υπόβαθρο μπορεί να οδηγήσει συγκεκριμένε ανισότητε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, πιο ηλικιωμένε ε, γυναίκε λένε ότι υπήρξε μικρότερη ζήτηση για αυτά, έστω και αν οι δεξιότητε εξελίχθηκαν με τον καιρό. Ή στην Αυστρία, ε, επίση, ε, υπήρξαν κάποιες διακρίσεις όσο προχωρούσε η ηλικία τους. Αν και οι διακρίσεις αυτές μπορούν να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο από χώρα σε χώρα. Ε, σε άλλες χώρες είναι ακόμα πιο τραβηγμένα τα στερεότυπα του φύλου. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, θα ήθελα να σε επισημάνω ορισμένου ε, παράγοντες κλειδί στα ΜΜΕ. Καταρχήν, οι άμεσες διακρίσεις. Ιδιαιτέρως στην Μάλτα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστρία και σε μικρότερο βαθμό στη Σουηδία άμεσες ε, διακρίσεις κατά το γυναικών είναι σημαντικό πρόβλημα στα ΜΜΕ. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουν να παλέψουν πιο σκληρά από τους άντρες για να έρθουν στο ίδιο επίπεδο αντιμετώπισης. Ε, μία γυναίκα είπε ότι δούλευε για ένα δημόσιο ραδιοφωνικό φορέα και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να έχει τις ίδιες αποδοχές με τους άντρες συναδέλφους. Ε, ε, και τελικά στιγματίστηκε γιατί προσπάθησε να επασπιστεί τα δικαιώματά της και ε, κατέβαλε ένα υψηλό τίμημα επειδή επέμενε στα δικαιώματά της. Όσον αφορά την κατανομή της εργασίας, πολλές φορές οι γυναίκες συστηματικά παραμελώνται ε, και δεν ε, προωθούνται στον ε, τομέα της οικονομικής ή πολιτικής δημοσιογραφίας ή ασχολούνται περισσότερο με τα πολιτιστικά. Τώρα, η παρενόχληση και αυτή ήταν ένα σημαντικό θέμα σε όλες τις χώρες που κάλυψε η έρευνα. Οι περισσότερες γυναίκες είχαν υποστεί παρενόχληση στη, στο χώρο εργασίας τους, δηλαδή ε, σεξουαλικές προτάσεις από πελάτες, συναδέλφους, managers και τους ε, ε διοκτήτες των ε, ΜΜΕ. Ε, σε ορισμένε χώρε εργασία η παρανόχληση δεν γινόταν ανεκτή. Σε, αλλού, σε, άλλα, άλλους χώρους ασκείτο συστηματικά. Όταν οι γυναίκες σε ορισμένες, ε, ορισμένες φορές οι γυναίκες ε, καλούνται να δημοσιοποιήσουν τις ε, περιπτώσεις παρενόχλησης. Η εκστατεία ε, η οποία έγινε περιλάμβανε ζητήματα ατιμορρησίας και αποσιώπησης και είχε σαν στόχο να αυξηθεί η συνειδητότητα της, ε, του φαινομένου και ανάγκη επαρκούς αντίδρασης. Ε, στην Αυστρία υπήρχε πιο συντηρητική ανταπόκριση στην εξαρτία αυτή, μη του, Εντό των ΜΜΕ και εκφράστηκαν κάποιες αντιρρήσεις λέγοντας ότι η εξαρτία αυτή είναι υπερβολική. Και πάντοτε να και στις γυναίκες το να αρνηθούν μια σεξουαλική πρόταση. Ε, βεβαίως... Ε, πολύ συχνά υπάρχουν ε, αρνητικές ε, επιπτώσεις αν μια γυναίκα προσπαθήσει να προωθήσει ιδέες περί ισότητας. Βεβαίως, από την εξαρτία και μετά, άρχισαν οι γυναίκες να δημοσιοποιούν τις, την περίπτωσή τους, απαιτώντας δικαιοσύνη. Φάνηκε ότι υπάρχει συστημική έλλειψη δικαιοσύνης, απόδοσης δικαιοσύνης στις περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν αρκετά ένδικα μέσα και πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι διάφορε πλευρέ στην περίπτωση τη παρενόχληση και τι είδου σύστημα πρέπει να ισχύει. Με τα ισχύοντα συστήματα μπορεί να διατηρηθεί η παρενόχληση χωρί πρόβλημα μακροχρόνια. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει πιο διαρκεί λύσει ιδίω για τι βιομηχανίε ε, των μέσων μαζική ενημέρωση, η διακριτική μεταχείριση και η παρενόχληση, παρά τι ε, σαφεί ευρωπαϊκέ και εθνικέ πολιτικέ, δεν λειτουργούν. Πολλέ φορέ όσοι δουλεύουν στα μέσα είναι πολύ ανταγωνιστικοί ω επαγγελματίε. Και πολλέ φορέ η εργασία freelance είναι πολύ συνηθισμένη στη δημοσιογραφία, στην τηλεοπτική παραγωγή. Γι' αυτό είναι και επισφαλή οι θέσει οι γυναίκες λοιπόν πολλές φορές, εάν ε, γίνουν αντιληπτές, εάν θεωρηθούν ταραξίες, ε, δυσκολεύουν την εξέβρεση εργασίας. Ο επισφαλής αυτός χαρακτήρας ε, στην δουλειά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει να κάνει και με το πόσο εύκολο να γίνονται τελικά ανεκτές αυτές οι συμπεριφορές. Οι γυναίκες στην πράξη, εφόσον υποστούν κακοποίηση παρενόχληση, δεν έχουν και κάποιο πραγματικό ενδικό μέσο το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και πολλές φορές έχουν την εντύπωση ότι αν αντιδράσουν μπορεί να χάσουν την καριέρα τους. Υπάρχει λοιπόν επίγουσα ανάγκη να αναλυφθεί δράση ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι κανόνες για την ίση μεταχείριση στην ε, εργασία, ιδίω για την ανισότητα, τη μισθολογική ανισότητα και την οικοποίηση, μπορεί να επιβληθούν οι σωστοί κανόνες με τους κατάλληλους μηχανισμούς ε, και τις δέουσες διαδικασίες ώστε τα ε, ένδικα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς να μην του κοστίσουν την καριέρα του. Αυτό και στον τομέα των μέσων και αλλού. Τώρα για την ε, συμμετοχή στον ε, χώρο εργασίας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις γυναίκες που έχουν παιδιά. Ε, όταν πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους ε, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα όπως εντοπίστηκε στην Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο χάρη να συνδυάσουν επαγγελματικό και οικογενειακό βίο. Οι, βίο. Οι εργοδότες φορές δεν θέλουν να πληρώσουν τη γονική άδεια ή την άδεια μετρότητα. Και όταν οι γυναίκε, ε, επειδή έχουν κάνει παιδιά, φύγουν για πολύ καιρό από τη δουλειά του, αντιμετωπίζουν σοβαρά μειονεκτήματα σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό νομικό. Και επίση λόγω τη ταχύτητα εξέλιξη τη τεχνολογία στον τομέα των μέσων. Κάθε χρόνο η τεχνολογία αλλάζει. Ό,τι συμβαίνει με την ε, με τις κάμερες λόγω χάρη, την συνδεξία, το editing, ε, από τι ειδήσει μέχρι την ψυχαγωγία και τη διαφήμιση τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Είναι λοιπόν δύσκολο να φύγει κανεί για πολύ καιρό από την ενεργοδράση δράση χωρί να πληρώσει τι συνέπειε. Επίσης τονίζεται ότι είναι τεράστια τα ωράρια εργασίας που απαιτούνται στα περισσότερα μέσα, 18 ώρες την ε, ημέρα. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει κανείς αρκετό χρόνο με την οικογένειά του και αυτό αφήνει πολλές γυναίκες, ιδίως όσες είναι υπεύθυνε ε, για την φροντίδα των παιδιών ή για την ε, δουλειά στο σπίτι, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν ικανοποιητικέ καριέρες. Απαιτούνται πολλές θυσίες από άλλους τομείς της δουλειάς τους. Αυτό έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογική τους υγεία. Τώρα να θέσω ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε συνολικά. Η διευρυμένη πρόσβαση στην μερική απασχόληση και την ευέλικτη απασχόληση είναι ένα τρόπο να υπάρξει εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου. Είναι μέρο των προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική ατζέντα. Είναι δύσκολο όμω να εφαρμοστεί με δίκαιο τρόπο, εκτό αν υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα που να τα προβλέπουν οι ίδιε οι εταιρείε και να τα ακολουθούν προσεκτικά οι μάνατζερ. Η αποτύπωση λοιπόν τη σημερινή εικόνα δείχνει ότι είναι πολλέ οι γυναίκε που προσλαμβάνονται για να δουλέψουν ε, σε θέσει μερική απασχόληση, αλλά τελικά τα συμβόλαια που του δίνονται καλύπτουν περισσότερε ώρε από ό,τι πραγματικά δουλεύουν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει επέκταση τη μερική απασχόληση στον τομέα των μέσων και οι γυναίκε να λαμβάνουν λιγότερα, μικρότερε αμοιβέ για το χρόνο που έχουν δουλέψει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά, διότι οι εταιρείε κοινωνία μπορεί να χρησιμοποιήσουν τους κανόνες για να βεβαιωθούν ότι οι γυναίκες ε, αξιοποιούνται στο επίση μπορεί να γίνει με τρόπο υπόγειο ή πλάγιο και να μην είναι φανερός ε, πολλές φορές είναι, ε, ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν την απόρριψη εργαζόμενων στον χώρο των ε, μέσων ενημέρωσης. Τελικά φαίνεται ότι Εάν δεν αναλυθούν ε, βήματα για να βεβαιωθούμε ότι καλύπτεται το μισθολογικό χάσμα ε, σε ομάδες και συνεδριάσεις, θα... εάν δεν αναλυθούν ε, βήματα για να βεβαιωθούμε ότι καλύπτεται το μισθολογικό χάσμα σε ομάδες και συνεδριάσεις, θα υπερέχουν πάντα οι άντρες. Άρα, αλλάζει και ο τρόπος επικοινωνίας. Οι φωνές που ακούγονται ε, περισσότερο και πιο δυνατά είναι αντρικές και οι διαφωνίες ε, παραγωνίζονται αμέσως ε, διότι εκφράζουν μια διαφορετική. Ακολουθηθούν οι δημιουργικές τους ιδέες ενώ οι γυναίκες εκφράζουν την άποψη ότι οι γυναίκες που εκφράζουν την άποψή τους ηχηρά μπορεί να κερδίσουν μια διαπάλη αλλά πολλές φορές θα τις ταυτίσουν με άντρε. Ε, υπάρχει λοιπόν πρόβλημα στην επικοινωνία, γιατί οι γυναίκε θεωρείται ότι πρέπει να εκφράζουν διακριτικά και όχι ανταγωνιστική στι εταιρείε και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Επίση, είναι πολύ σημαντικό ε, να δούμε το χώρο εργασία, τον τόπο εργασία και την διαδικασία λήψη όχι και βλέπουμε ότι πολλέ φορέ τα δυσάρεστα φαινόμενα λαμβάνουν ε, χώρα το βράδυ. Όταν κάποιοι βγαίνουν για ποτό για να τα πούνε μετά τη δουλειά, τότε που οι γυναίκε πολλέ φορέ πρέπει να γυρίσουν σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά και δεν μπορούν να ακολουθήσουν a η διαρκής λοιπόν ε, διακριτική μεταχείριση, η κακοποίηση μπορεί να ε, έρθει σε αντίθεση με την ε, εκκλήση των καθηκόντων της μητέρας που μπορεί να έχει μια γυναίκα ή την όλη νοοτροπία, τον τρόπο που επικοινωνούν οι άντρες. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το περιεχόμενο της ελευθερίας της έκφρασης. Όμως, ένα σύνολο κανόνων μπορεί να δημιουργήσει και το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να υπάρξει αποστοχώρηση στις αξίε. Πάντως, η παρουσία των γυναικών είναι σαφώς ε, οπισθοδρομική, ε, είναι στερεοτυπική. Οι κυρώσεις δεν χρησιμοποιούνται, τα πρόστιμα δεν ε, επιβάλλονται. Παρόλο που βλέπουμε νέε οδηγίε να αναδύονται, οι ρυθμιστέ, οι νομοθέτε θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να υπάρξει κατάλληλο συντονισμό για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων. Παρόλο που υπάρχουν λοιπόν οδηγίες και κανόνες, οι περισσότεροι από όσου ε, ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας από τη Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν τους γνώριζαν καν. Ε, στα ψηφιακά επίσης μέσα υπάρχουν ε, και κίνδυνοι και ευκαιρίες, όπως συζητήσαμε σήμερα και βλέπουμε να ε, υπάρχει διαρκής αναγνώριση του ότι μπορεί να υπάρξει περιεχόμενο με τάσεις διακριτικής μεταχείρισης και σε διάφορες επιγραμμικές πλατφόρμες. Είναι διαφορετικό λοιπόν Πρέπει κανεί να κάνει τη σωστή διάκριση μεταξύ τη προσφορά ε, περιεχομένου και ε, του κατά πόσον κάποιο πέφτει θύμα του περιεχομένου αυτού. Ε, η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή δημοσιογραφία είναι ένα τομέα που προοδεύει γοργά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι αν αυτό είναι το μέλλον τη δημοσιογραφία, οι γυναίκε δεν θα μείνουν απ' έξω. Οπότε θα ήταν θετικό να έχουμε προσπάθειες που αποβλέπουν στην αύξηση τη συμμετοχή των γυναικών, ιδιαίτερα στην κατάρτιση σε αυτό το τομέα. Σχετικά με περιπτώσεις διακρίσεων και οχλήσεων που συνεχίζονται παρά την ύπαρξη νομοθεσιών. Θα πρέπει να εντοπίσουμε άμεσο τα θέματα που συνεχίζονται παρά την ύπαρξη νομοθεσιών. Θα πρέπει να εντοπίσουμε άμεσο τα θέματα γυναίκε τη δυνατότητα πραγματικής προσφυγής χωρίς αυτή δηλαδή να επιφέρει κινδύνους στη σταδιοδρομία τους. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι εσωτερικές πολιτικές είναι διαφανείς, είναι ισότιμες και ότι είναι δίκαιες. Και εδώ θα πρέπει όμως να, προωθήσουμε, να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις αμοιβέ και αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια προϋπόθεση και μάλιστα η διαφάνεια αυτή να επεκταθεί σε όλους τους, σε όλες ε, κλίμακες και στα κριτήριά τους. Η, η κανονικοποίηση της ημιαπασχόλησης είναι πρόσδεκτη, όμως θα πρέπει να πετύχουμε το σωστό συντονισμό στον χώρο εργασία, ώστε να διασφαλίσουμε στους ημιαπασχολούμενους την σωστή διάρκεια εργασίας στη σωστή διάρκεια πρέπει να διευρυνθούν, να επεκταθούν θα πρέπει να εντάξουμε εδώ και δεξιότητες που επιτρέπουν αμοιβέ που θα περιλαμβάνουν γονική και μητρική άδεια και επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιστροφή των γυναικών μετά από τη μητρότητα. Στα ΜΜΕ ε, η επιστροφή αφού γίνει πρέπει να συνοδεύεται από κάποια κατάρτιση που, θα έχουν χαρακτήρα εξισωτισμού και πρέπει εδώ να μπλέξουμε και παρικά όργανα και οργανισμούς στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε και οι επιχειρήσεις να γίνουν και αυτές πιο προσεκτικές όσον αφορά τα θέματα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον τομέα του ΜΜΕ θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο. You know, uh, Όπως ξέρετε, προετοιμάσαμε την έκθεσή μας πριν από την. Λοιπόν, ενδιαφέροντα τα ευρήματά σας και η μελέτη σαν αναπερίπτωση για τις χώρες μέλη. Πρέπει κάπου να τα διαβάσω προσεκτικά γιατί όλα αυτά είναι νέα στοιχεία για μένα όσον αφορά τη δημοσίευσή σας. Έχω λοιπόν κάποια ποια είναι αυτά τα νέα εργαλεία πολέμησης της ανισότητας στο χώρο εργασίας στα ΜΜΕ. Δηλαδή, τι μπορείτε αυτή τη στιγμή να προτείνετε ως κάτι χρήσιμο και απτό εργαλείο. Υπόψη σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Tack så mycket Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την ε, που μου δίνετε λόγο και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ενδιαφέρουσα εισηγήσή τη. Το σημείο αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Yeah. Των γυναικών. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το σημείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι συμβαδίζει με όλα αυτά που αναφέρει και η έκθεση. Αλλά νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αυτό το πράγμα. Έχουμε ε, τα φαινόμενα σεξισμού που και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Οι γυναίκες νομίζω ότι θέλουν να εργάζονται. Αντίθετα, μας απασχολούν περισσότερο οι τρόποι πλήρους εργασίας, οι μορφές πλήρους εργασίας για τις γυναίκες, ώστε αυτές να είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε αυτά τα αιτήματα ε, για τα οποία μιλήσατε προηγουμένως, ε, από ποιες χώρες προέρχονται, δηλαδή αυτή, αυτό το αίτημα που υπάρχει, το γενικό για μια απασχόληση, από πού προέρχεται. Ευχαριστώ πολύ την συγγήτρια για την εισήγησή της. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία μας είχε ρωτήσει κάτι σε σχέση με την οδηγία που αφορά μορφές διάκρισης, μίσους, παρότρησης βίας κλπ. Σχέση με αυτές τις δομές που προβλέπει η έκθεσή σας, αυτές οι ίδιες από μόνες τους αυτές τις δομές αποτελέσουν εγγύηση, εξάλληψης, ε, διακρίσεων, μίσους κτλ. Δηλαδή θα έχουμε ένα ενιαίο όπλο, ένα ενιαίο εργαλείο για την αλλαγή των δομών, κάτι το οποίο μου φαίνεται δύσκολο. Θα πρέπει να δούμε το θέμα σφαιρικότερα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γενικότερα, όχι μόνο για τα οπτικοακουστικά ή τα ΜΜΕ, αλλά γενικότερα. Ε, οι ποσοστώσει. Από ό,τι ξέρω, στην Πορτογαλία υπάρχει κάτι τέτοιο, προβλέπεται και είναι αποτελεσματικό έχει νομοθετήσει το μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε υψηλότερο επίπεδο. Επίσης, να καταλήξω λέγοντας το εξής. Τι γίνεται με την όχληση και κατά πόσο οι γυναίκες την αναγνωρίζουν. Εκτός μικροφώνου, να ακούμε Χριστό. να um, Θα απαντήσω τις ερωτήσεις σας και θα επανέλθω και στα εργαλεία για την εξασφάλιση περισσότερης ισότητας στα ΜΜΕ. Συμφωνώ απολύτως ότι αυτές οι ανισότητες είναι αλληλένδετες ε, και χρειάζεται βεβαίως μια περιεκτική στρατηγική